μισή. Κυρίε και κύριοι, επόμενη συνεδρίαση αύριο 12 Ιουνίου 2013 στις 8.30 έως τις 2 το απόγευμα. Έχει δημοσιευτεί η ημερήσια διάταξη και είναι διατίθεται στον ιστοτόπο του Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση λίγη.